morning to everybody. Our president uh, is a little bit busy. Our chairwoman is a little bit uh, busy right. Είναι απασχολημένη η πρόεδρος μας, άρα ε, θα αφήσουμε ε, τα σχετικά με την συνάντηση των συντονιστών και τα όσα αποφασίστηκαν για όταν θα έρθει. Ε, συμφωνήσαμε ότι ο κ. Μποστινάρου μπορεί να μας εξηγήσει τη γνωμοδότησή του περί βιοπικιλότητας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το έγγραφο εργασίας με την ονοματότησή μας και με τα σχετικά από, προηγούμενες, ε, από προηγούμενα έτη βρίσκεται υποσύνταξη και θα σας, το, θα σας το διαβιβάσω στην επόμενη συνεδρίαση. Για λίγα λεπτά θα σας πω ποια είναι τα βασικότερα του σχεδίου εκθέσεως καθώς και τα συμπεράσματα τα οποία εμπνέονται από τις προηγούμενες δραστηριότητές μας, από τις εκθέσεις και κυρίως από τις αναφορές που έχουμε λάβει από πολίτες ε, των, ε, της Ενωμένης Ευρώπης, ε, κυρίως για θέματα περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας. Γιατί η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να αναμειχθεί στο θέμα αυτό. Κατά τη γνώμη μου, είναι σωστό, διότι στην Επιτροπή Αναφορών Κατ' επανάληψη έχουν αποστείλει και μεγάλο αριθμό αναφορών οι πολίτες σχετικά με τη βιοπικιλότητα. Έτσι λοιπόν έχουμε και τεχνογνωσία του θέματος, έχουμε και βαθύτερη γνώση της βιοπικιλότητας και του τρόπου με τον οποίο ε, θίγεται η βιοπικιλότητα και εθίγει τελευταία από διάφορα κενά στις διαδικασίες εφαρμογής αλλά και από την ασθενή εποπτεία και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τις χώρες μέλη. Σημαντικός αριθμός αναφορών για το περιβάλλον προέρχονται από όλες τις χώρες μέλη αναφέρονται σε μία εφαρμογή οδηγιών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής νομοθεσίας και των προγραμμάτων για την αναχέτηση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Θα περάσω τώρα στο σχέδιο δράσης που υποτίθεται ότι ε, θέλει να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέχρι το 2010. Το σχέδιο απέτυχε και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την αποτυχία και λέει ότι είναι πολύ απίθανο να επιτευθεί ο στόχος της ε, ανακοπής της απώλειας βιοποικιλότητας του 2010. Αναμένοντας νέο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το 2010, εγώ άκουσα ότι ολοκληρώθηκε η σύνταξη του σχεδίου και διαβιβάστηκε το σχέδιο ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. 50% των ειδών, ε, σημαντικό ποσοστό των οικοτόπων που ωστόσο προστατεύονται από την οδηγία οικοτόπων, ε, βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση. Πάνω από 40% των πουλιών, που, των ειδών των πουλιών δηλαδή, ε, βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση από άποψη ε, διατήρησης. Όλο και περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις λόγω της ανάπτυξης η απώλεια βιοπικιλότητας και οικοσυστημάτων, η διατήρησή τους μάλλον είναι σημαντική για την ευημερία όλων. Σημαντικές είναι οι οδηγίες περί προστασίας των πουλιών και των ε, οικοτόπων, Natura 2000 και προστατευόμενες περιοχές, 17% της ευρωπαϊκής επικράτειας καλύπτεται τώρα από αυτές τις σημαντικές οδηγίες. Εάν όμως αυτό το ποσοστό καλύπτεται από το σχέδιο Natura 2000 και προστατευόμενες περιοχές, δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τους άλλους κανονισμούς και κανόνες, όπως για την μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον, την οδηγία προστασίας των νερών, καθώς και το νομικό οπλοστάσιο για την διαχείριση των δασών της γεωργίας, της Αλίας και των ε, υδατοκαλλιεργιών. Κάποια πρόοδος έχει γίνει, όπως δείχνουν ωστόσο οι δείκτες. Ο στόχος της Biodiversity 2000 δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Η κλίμακα απώλειας βιοπικιλότητας σημαίνει ότι απαιτείται άμεση ανάληψη δράσης. Τι μπορούμε τώρα να αμεμφθούμε. Πρώτα, έλλειψη ε, σαφήνειας, καθώς και ασάφεια ορισμένων διατάξεων μέσα στις ίδιες τους κανονισμούς της Ένωσης. Μη ξεκάθαρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και, και ε, ελλειπής εφαρμογή των ε, κανονισμών. Εάν συνεχίσουμε έτσι, υποσκάπτουμε την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος Πράγματι, παρόλες τις αρχές της προφύλαξης και της αναλογικότητας, οι δημόσιες αρχές πάντοτε βάζουν τις δικές τους στενές οικονομικές προτεραιότητες πάνω από την ανάγκη διατήρησης των ειδών και ιδίως όταν εμπλέκονται και σημαντικά οικονομικά λόμπι, μεγάλες επιχειρήσεις και μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ξεκολουθούμε να μην έχουμε σημεία αναφοράς για σύγκριση. Χρειαζόμαστε συνεπές monitoring για να καταδεικνύουμε τις επιπτώσεις και για να προτείνουμε καλύτερες λύσεις. Ποιες είναι οι προκλήσεις τώρα για την εφαρμογή και την βελτίωση της ε, παρούσας κατάστασης. Πρώτα, υπάρχουν καθυστερήσεις για την ε, εφαρμογή στο 17% της επικράτειας. Δεύτερο, ελλειπής διαχείριση. Μελέτη, μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον και στατικές μελέτες οι οποίες σπάνια είναι ικανοποιητικέ σε σχέση με την προστασία της βιοπικιλότητας. Η δική μου σύσταση θα είναι στην έκθεσή μου να αναφέρουμε επίσης την ανάγκη πιστοποίησης των επιχειρήσεων εκείνων που κάνουν μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για τον απλό λόγο ότι συχνά, τόσο συχνά, οι μεγάλες επιχειρήσεις προτιμούν να πληρώνουν λιγότερα χρήματα για τις μελέτες και να αρχίζουν αμέσως τα έργα και αυτά έχουν βέβαια τρομερές συνέπειες στην ε, βιοπικιλότητα. Υπάρχει ανάγκη και περαιτέρω πρόοδου ώστε οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υποτίθεται ότι γίνονται συστηματικά για περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν οι χώρες μέλη για την αποφυγή των ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. υπάρχει και μεγάλη απόσταση μεταξύ μέτρων και εφαρμογή των μέτρων από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη στιγμή δηλαδή όπου ε, ειδοποιείται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι ότου ε, αντιδράσει και μέχρι ότου τα μέτρα ε, αρχίσουν να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται από τις χώρες μέλη υπάρχει τέτοια μεγάλη καθυστέρηση ώστε προκαλούνται σημαντικές ζημίες. Θα πρέπει να περιορίσουμε τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης και των χωρών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι θεμοί τους αφήνουμε ανοιχτές πόρτες και παράθυρα να μας προσφέρουν αδύναμες εξηγήσει για ποιο λόγο καταραίει η βιοπικιλότητα. Και έτσι δεν μπορούμε να ανατρέψουμε την αρνητική αυτή κατάσταση. Ο χρόνος Αντίδραση στην, στην ε, καταστροφή της φύσης των εθνικών αρχών είναι πάρα πολύ σημαντικός, πάρα πολύ μεγάλος. Και όχι μάλιστα μόνο στι νέε χώρες μέλη, αλλά και στις παλιέ. Σπανιότατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά θέματα επιτόπου και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη πλήρων απόψεων σε σχέση με τις αναφορές οι οποίες έχουν διαβιβαστεί σε αυτήν. Τόσο συχνά βλέπουμε εδώ στην Επιτροπή Αναφορών την πραγματικότητα ότι δηλαδή οι επίσημες απαντήσεις που λαμβάνουμε και από τις χώρες μέλη και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τόσο ασαφείς. Στερούνται συνέπεια, ώστε κάτι πρέπει να αλλάξει. Η Επιτροπή Αναφορών πρέπει κάτι να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή. Εν συμπεράσματι στο κεφάλαιο αυτό σημειώνω τα προβλήματα της διαχείρισης, χρηματοδότησης, εφαρμογής και αξιολόγησης. Χρειαζόμαστε επίσης πιο φιλόδοξους στόχους και περισσότερη δέσμευση. Πρώτα, η οδηγία περί μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι κυρίως διαδικαστικού χαρακτήρα και είναι ασθενής και στην πραγματική της εφαρμογή και για ε, οικοσυστήματα όπου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα δεν αποδίδει τον πραγματικό της στόχο, δηλαδή να διασφαλίζει ότι το φυσικό περιβάλλον αλλά επίσης και η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά να προστατεύεται εύλογα από την καταστροφή που προκύπτει από την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να ενισχύσουμε επίσης την οδηγία ώστε να επιτρέπει ταχύτερη αντίδραση και μάλιστα και με έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας και της Επιτροπής Αναφορών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος για να βελτιωθεί η τρέχουσα νομοθεσία. Άλλα θέματα τα οποία, ε, για τα οποία έδωσε έμπνευση η μελέτη που κάναμε το φθινόπωρο. Η διάσταση της βιοποικιλότητας που σήμερα ασχολούμαστε με τη βιοπικιλότητα σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Αλλά, αλλά υπάρχουν προβλήματα και διαμεθοριακού χαρακτήρα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε για να βελτιώσουμε και νομικά την διαμεθοριακή διαχείριση της ε, διάστασης της βιοπικιλότητας. Εν προκειμένου και, συμπληρώνω, και ολοκληρώνω αμέσω, εν προκειμένου θα σας προτείνω να ζητήσουμε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλουν στις θεσμικές, θεσμοποιημένες μας σχέσεις με τους γείτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νομικό προστάσιο που διαθέτουμε ώστε να καταστεί δεσμευτικό και για τις ε, γειτονικέ αυτές χώρες. Διότι όταν τα προβλήματα που έχουν σχέση με την μείωση της βιοποικιλότητας προέρχονται Βεβαίω έχουμε και εμείς αδυναμίες και προβλήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν τα προβλήματα, για παράδειγμα ρήπανση ή μεγάλα έργα υποδομών, προέρχονται από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουμε νομικό προστάσιο για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και να διορθώσουμε το πρόβλημα. Η έκκλησή μου προς εσάς και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι να εντάξουμε στις θεσμοποιημένες μας σχέσεις και το νομικό προστάσιο που είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά. Για παράδειγμα το πρόβλημα της ενέργειας, της, ενέργειας, το, της διαχείρισης των νερών και ούτω καθεξής. Έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της ε, διατήρησης της βιοποικιλότητας. Εν τέλει, το συμπέρασμά μου νομίζω είναι πολύ σημαντικό χρειάζεται να ασκήσουμε πίεση για πλήρη εφαρμογή τη τρέχουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλλαγέ στην νομοθεσία αυτή, βελτιώσει είναι απαραίτητες. Αυτό που χρειαζόμαστε όμω παραπάνω απ' όλα είναι να φροντίσουμε για την πλήρη εφαρμογή της από τις χώρες μέλη, καθώς επίσης και στενότερη παρακολούθηση, monitoring από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν μια χώρα μέλος δεν εφαρμόζει την νομοθεσία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ και θα σας προσκαλέσω όλους να συμβάλλετε με τις ιδέες σας. Σας υπόσχομαι ότι θα περιλάβω όλες τις προτάσεις σας, τροπολογίες, ιδέες κλπ. Και μετά θα εργαστούμε όλοι μαζί επί της τελικής μορφής του εγγράφου. Σας ευχαριστώ πάντως για την προσοχή σας και την επόμενη εβδομάδα θα σας διανύμω το πρώτο μου σχέδιο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρο. Ξαναδίδω βεβαίω τα ενία της διεύθυνση της συζήτησης στην ε, Πρόεδρο. Λόγω στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Χονσουά Κρεμέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε ξανάρθει στην Επιτροπή Αναφορών, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την έκθεση. Γνωρίζουμε την κατάσταση, η οποία δεν είναι λαμπρή. Και ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα φτάσει στο στόχο της ε, να ανατρέψει την, την προβληματική κατάσταση για τη βιοπικιλότητα μέχρι μέχρι το 2010. Η Κομισιόν θα παρουσιάσει μια νέα ανακοίνωση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη χρονιά που είναι η χρονιά της βιοπικιλότητας για να ενδυναμώσουμε τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της βιοπικιλότητας το οποίο πέρα από την κλιματική αλλαγή είναι το νούμερο δύο μείζον πρόβλημα. Ε, ο κύριος Ποστινάρου ανέφερε τα προβλήματα, τα γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι εδώ στην Επιτροπή Αναφορών διάφορες αναφορές ε, υπάρχουν για παραβιάσεις τις οποίες διερευνά η Επιτροπή και είναι οι περισσότερες στον αριθμό. Είναι ο πρωταθλητής της υποθέσης που παρακολουθεί η Κομισιόν. Συχνά υπάρχουν παράπονα γιατί δεν υπάρχουν είτε ενημέρωση είτε δεν λαμβάνονται αποφάσεις. Αυτό ίσως να οφείλεται και στις αόριστες πληροφορίες που λαμβάνουμε. Τότε στρεφόμαστε εκ νέου προς τους αναφέροντες και ζητάμε νέες πληροφορίες. Ε, και ακριβώς εκεί ξοδεύουμε πάρα, πολλές, πάρα πολλούς πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλοί συναδελφοί μου παίρνουν τον χρόνο τους διερευνώντα αυτά τα πράγματα. Ε, προχωρούμε σε δράση ε, και επισήμως σε πολλές περιπτώσεις, το ξέρετε εσείς, στα θέματα περιβάλλοντος. Παραδείγματο χάρη για τη Βία Μπάλτικα. Εκεί σταματήσαμε να ανακόψουμε μια πορεία καταστροφική ε, και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δρούμε προληπτικά τώρα. Έχουμε δημιουργήσει ένα μοναδικό δίκτυο για την ε, προστασία κάποιων ε, φυσικών περιοχών, που δεν είναι απλές φυσικές περιοχές, είναι 25.000 και είναι, θέλουμε να τις βοηθήσουμε να διατηρηθούν βιώσιμα. Υπάρχει αυτό το δίκτυο λοιπόν, το οποίο είναι φημισμένο σε όλο τον κόσμο και προσπαθούμε να υπάρξει σωστή διαχείριση. Και νομίζω ότι αυτό, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Τώρα, από την πλευρά των κρατών μελών ε, υπάρχει υποχρέωση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης και διατήρησης, να εντοπίσουν στόχους συντήρησης και διατήρησης για να υλοποιήσουμε τον κοινό στόχο να επαναφέρουμε κάποιους χώρους σε καλή κατάσταση διατήρησης. Ξέρετε, το αναφέρετε κι εσείς, ότι πολλά τέτοια, τέτοιες περιοχές είναι σε κακή κατάσταση. Οι εκθέσεις του άρθρου 17, το 50-60% των οικοτόπων είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Νομίζω ότι αν καταφέρουμε να προσεγγίσουμε το θέμα από την πλευρά της διαχείρισης ε, και της χρηματοδότησης θα, κάνουμε, θα σημειώσουμε πρόοδο. Το αναφέρατε και εσείς στην εκθεσή σας, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Έχουμε κάποια εργαλεία. Έχουμε αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Ε, έχουμε προβλέψει 20 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για την φύση και τη βιοποικιλότητα. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Βέβαια τώρα το μπαλάκι είναι στα κράτη-μέλη. Εμείς δεν έχουμε άλλη επιρροή. Επηρεάζουμε από πλευράς μας κάποια προγράμματα, κάνουμε ό,τι μπορούμε και στο περιβάλλον προσπαθούμε να παρισφρήσει και η έννοια της του φυσικού περιβάλλοντος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά αν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν και αυτά ό,τι μπορούν και αν ο οικονομικός ε, τομέας, οι οικονομικοί φορείς δεν κατανοήσουν ότι η ανάπτυξη των ε, βιομηχανιών τους μπορεί να πετύχει μόνο αν είναι βιώσιμη από φυσικής και περιβαλλοντικής ε, πλευράς, μόνο τότε θα υπάρξει επιτυχία. Μια, προωθούμε μια εκστρατεία αυτή τη χρονιά του το 2010 για να προωθήσουμε τη βιοπικιλότητα. Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες της Κομισιόν τα τελευταία χρόνια για να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για την υπάρχουσα νομοθεσία και είμαστε πεπισμένοι ότι η οδηγία για τους οικοτόπους είναι ένα θαυμάσιο και μοντέρνο εργαλείο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να γίνει κατανοητό και έχουμε γι' αυτό κατευθυντήριες γραμμές. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε ξεκινήσει το, με τις τομεακές κατευθυντήριες γραμμές που είναι τομείς που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι όπω τα λιμάνια, ε, οι μη εξορυκτικές βιομηχανίε, ε, το δέλτα των ποταμών, οι εσωτερικέ υδάτινε οδοί και προσπαθούμε ε, να βρούμε εταίρους σε, αυτό το, σε αυτή την προσπάθεια στα πλαίσια του Natura 2000. Μιλάμε για τομείς που θα πρέπει να εμπλακούν ε, και να αναπτυχθούν με έναν τρόπο ώστε να γίνει καλύτερο το περιβάλλον. Σε πολλά προγράμματα είναι εύκολο να σημειωθούν θετικά βήματα. Όχι μόνο να αποφευθεί η επιδείνωση, αλλά να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Η οδηγία για του οικοτόπου βασίζεται σε αυτήν την προσέγγιση και η λέξη, α, υπάρχει, υπάρχει η λέξη κλειδί επιδείνωση και αποκατάσταση ε, μέσω της αποζημίωσης. Καλά είναι αυτά αλλά είναι το ελάχιστο. Θέλουμε τα προγράμματα τα οποία αναπτύσσονται, αλλά να μην επιδεινώνουν την κατάσταση, αλλά ε, συνεργάζονται και αυτά για την υλοποίηση των στόχων του Natura 2000. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν στην ε, ισχύουσα νομοθεσία, λοιπόν. Και θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο για να πει εντάχει δύο λόγια για το έτος αυτό της βιοποικιλότητας. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Απλά και μόνο θα ήθελα να ενημερώσω το Κοινοβούλιο για τα, επόμενα βήματα ω προ την ανάπτυξη πολιτική. Όπω ε, είπε και η Πρόεδρο, η αξιολόγηση η οποία δημοσιεύθηκε στο τέλος του 2008 ήταν ενδιάμεση αξιολόγηση και με βάση αυτή τη συγκεκριμένη αξιολόγηση η Επιτροπή εργάστηκε ε, προ την κατεύθυνση μια ανακοίνωση που ανακρύφθηκε την περασμένη εβδομάδα στις 19 Ιανουαρίου και όπου αναφέρεται το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέχρι το 2015 και εκεί συμπεριλαμβάνονται επιλογές για ενδιάμεσους βασικούς ε, στόχους ε, που θα επιτευχθούν μέχρι το 2020. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα φιλοδοξίας και εδώ ελπίζουμε να υπάρξει ένα συνολικά ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Η πολιτική συζήτηση έχει τώρα ξεκινήσει. Έγινε αυτή η υψηλού επίπεδου συνδιάσκεψη στη Μαδρίτη την Τρίτη και Τετάρτη, ε, χτες και προχτές αυτήν την εβδομάδα, και όπου η Ισπανική Προεδρία τόνισε τη σημασία αυτού του ζητήματος και την αποφασιστικότητά της να υπάρξουν κάποια συμπεράσματα του Συμβουλίου το Μάρτιο τα οποία θα εγκριθούν και από το Ευρωπαϊκό το Συμβούλιο Κορυφής το Ιαρινό. Αυτές ε, είναι ε, οι απόψεις της Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική ε, μετά το 2010, μια πλήρη στρατηγική, συνολική στρατηγική επί του θέματος που ελπίζουμε να εγκρίνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου και εκεί έχουμε λάβει ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη για μια ε, βασική ε, γραμμή εκκίνησης, καθώς επίσης και τη σημασία των δικτών με τους οποίους θα παρακολουθήσουμε την πρόοδο ή την έλλειψη πρόοδου ε, μέχρι το 2020 και υποβολή έκθεση στο Κοινοβούλιο σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Επίσης, η Επιτροπή μέχρι το τέλος του 2010 θα δώσει τον πρώτο χάρτη των υπηρεσιών οικοσυστημάτων ε, στην Ευρώπη. Γιατί η βιοπικιλότητα δεν έχει να κάνει μόνο με την προστασία των ειδών και των οικοσυστημάτων, αλλά έχει να κάνει και με την παροχή των υπηρεσιών σε επίπεδο αποθήκευση ε, και δέσμευση του άνθρακα κτλ. Γιατί και όλα ε, αυτά τα στοιχεία μπορούν να έχουν άμεση σχέση με την οικονομία μας. Ελπίζω λοιπόν να καταλάβετε κι εσείς και να σας καθησυχάσαμε και να μας βοηθήσετε έτσι ώστε να εγκρίνουμε ένα ισχυρό φιλόδοξο στόχο, ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο να ενισχύσει και τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή γιατί θα έχουμε και την συνδιάσκεψη των μερών την ε, δέκατη, ε, την επόμενη, όπου πραγματικά θέλουμε να έχουμε ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία. Αυτά όσον αφορά ε, τις προσεχείς εξελίξεις. Ε, ναι, ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Μποστινάρου. Ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Είναι σαφές ότι όσον αφορά την έκθεση αυτή πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση. Λαμβάνοντας υπόψη ε, το χρονοδιάγραμμα ε, της Επιτροπής, είχαμε συμφωνήσει να ανοίξουμε τη συζήτηση, να αρχίσει η συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση. Δεν ξέρω τώρα, ε, αν θέλετε κυρία Όκεν να τοποθετηθείτε επί της ουσίας, οι παρεμβάσεις προγραμματίζονται για την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Ναι, πολύ σύντομο. Θα είναι πάρα πολύ σύντομη. Απλά και μόνο ήθελα να πω ότι το όραμα είναι μια ωραία λέξη. Αν όμως τα οράματα και οι ωραίες λέξεις μας έσωζαν, θα είχαμε ήδη σωθεί. Ε, γι' αυτό με φοβίζει τώρα αυτό το μήνυμα που ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί έχουμε νομοθεσία. Έχουμε τις δύο οδηγίες και είναι καλή. Πολύ καλή μάλιστα. Αλλά δεν εφαρμόζεται. Και δεν εφαρμόζεται ούτε από τα κράτη-μέλη, ούτε από την Επιτροπή. Και γι' αυτό με φοβίζει το όλο ζήτημα. Όταν ο Μπαρόζο είπε ότι θα υπάρξει αναθεώρηση, και ξέρουμε τι γίνεται στην Πορτογαλία. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά τρομοκρατήθηκα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει βελτίωση και του χειρισμού αυτής της υπόθεσης. Γιατί... Για δείτε την έκθεση που είχαμε πριν από λίγου μήνε που αφορούσε την οδηγία για την βιοποικιλότητα. Ε, δεν ξέρω. Ε, είναι ιδιαίτερα λυπηρή αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν, τι να πω. Βεβαίω όλοι θα βοηθήσουμε την Επιτροπή για να, για να έχουμε σωστή νομοθεσία, αλλά δεν είναι το πρόβλημα η νομοθεσία. Η πρακτική είναι το πρόβλημα. Just a small Μία σύντομη παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μποστινάρου. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι χαίρομαι με τις εξηγήσεις και τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις της Επιτροπής, αλλά υπάρχει εδώ μια επιφυλεκτικότητα, όχι μόνο σαν αφορά την πλήρη ε, εφαρμογή και υλοποίηση των υφιστάμενων κανόνων, αλλά σε δύο σημαντικές περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά ε, την ε, αναφορά ε, για το ρεύμα του κόλπου, για το North Stream. Και εκεί είχαμε πει ότι θα υπάρξει περιβαλλοντολογική αξιολόγηση όσον αφορά το θέμα αυτό, μια πολύ σημαντική αναφορά. Σήμερα φτάσαμε στο 2010, είναι Φεβρουάριος σχεδόν, αλλά κανένας δεν έχει πάρει κάποιες πληροφορίες από την Επιτροπή. για το ε, γεγονός ότι αυτή ε, η έκθεση είναι η καλύτερη λύση για τη διαφύλαξη της ε, Και όταν συζητήσαμε τη στρατηγική για την Βαλτική θάλασσα, μας είπε η ίδια Επιτροπή και ε, πρόσωπος της Σουηδίας, της Σουηδικής Προεδρίας, Ακούσαμε λοιπόν ότι η βαλτική ε, στρατηγική είναι συνολική, δεν υπάρχει χώρος για τη Ρωσία. Το καταλαβαίνω ότι η Ρωσία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ότι ε, ο αγωγός ε, Nord Stream είναι ένα εμπορικό ζήτημα το οποίο δεν εντάσσεται στρατηγική. Αν κάνουμε το ίδιο και με τη στρατηγική του Δούναβη και μετά για τη στρατηγική του Εύξηνου Πόντου, ε, και όταν ε, θα εξετάζονται τα διάφορα σχέδια μόνο ε, ε ως εμπορικά ζητήματα και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τεράστιες εταιρείες, πολυεθνικές εταιρείες. Τότε θα αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για το τι γίνεται στη φύση και γιατί έχουμε τέτοια απώλεια βιοποικιλότητας. Χρειαζόμαστε όμως μια συνολική και δεσμευτική λύση για την προστασία της βιοποικιλότητας γιατί διαφορετικά όλα αυτά είναι ευσεβείς πόθη. Και εμείς ε, δεν θέλουμε ευσεβείς πόθους και ευχές. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Ε, θέλουμε λοιπόν στην επόμενη συνεδρίαση, όταν θα αρχίσουμε τη συζήτηση και με τα μέλη της Επιτροπής, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει πιο συγκεκριμένες διασαφηνήσεις. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά ε, το στάδιο υλοποίησης των οδηγιών και γιατί ορισμένα σημεία της νομοθεσίας, παρά το γεγονός ότι είναι πλήρης, ε, δεν εφαρμόζονται. Και δεύτερον, γιατί εμείς δεν έχουμε πληροφορίες ε, για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Τι έγινε. Και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των αναφορών που έχουμε και που αφορούν το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα, το οποίο συζητάμε και σήμερα μέσα από την έκθεση του κυρίου Μποστινάρου. Να πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, στα δύο επόμενα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε αυτές τις 16 που βρίσκω, αναφορές βρίσκονται στα επόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 17 και 18. Ε, ομαδοποιήσαμε αυτές τις αναφορές γιατί ε, ε, αφορούν ένα κοινό θέμα γενικά. Δηλαδή πιο συγκεκριμένα το θέμα της επίγουσας ανάγκης από άποψη περιβάλλοντος στην Καμπανία. Πολλές αναφορές αφορούν την ε, συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή της Καμπανίας Άλλες αναφορές ε, καταγγέλουν ε, την, ε, ε, τις επιζήμιες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, συνέπεια της μη ορθής διαχείρισης των δομών που ασχολούνται με την διάθεση και διαχείριση των αποβλήτων στην Καμπανία, Ήδη έχουμε εργαστεί ε, και εργαστήκαμε στην ε, ε, συνεδρίαση την 1η Δεκεμβρίου, ακούσαμε τους αναφέροντες. Στο τέλος της συζήτησης και αφού ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαμε πει ότι θα ζητήσουμε, θα καλέσουμε τι εθνικέ εκπροσώπου των Εθνικών Αρχών και, των, ε, και της τοπικής αυτοδιοίκηση, δηλαδή και τη ιταλική κυβέρνηση και τη περιοχή τη καμπανία, για να δούμε πού βρισκόμαστε όσον αφορά την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει δράση επαλήθευση τη κατάσταση στην περιοχή της ε, Καμπανίας υπήρξαν, υπήρξε διαπίστωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίου και γι' αυτό ξεκίνησε διαδικασία παράβασης κατά της ε, Ιταλίας στην περιοχή της ε, Καμπανίας, η οποία και αυτή τη στιγμή το ζήτημα βρίσκεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην τελευταία συνεδρίασή μας επανέλαβε μας επανέλαβε ότι η δράση ε, έρευνας και επαλήθευσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Εξετάζεται το τι γίνεται μετά από τις νέες πρωτοβουλίες ε, που αναλύθηκαν σε τοπικό επίπεδο. Εξετάζεται λοιπόν η δυνατότητα ε, αποκατάστασης του θέματο και το κατά πόσο δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει για άλλη μια φορά η διάθεση και η χρησιμοποίηση κοινοτικών πόρων. Λοιπόν, να δώσουμε πρώτο το λόγο στον καθηγητή Άνταμ ο οποίο είναι ε, υπεύθυνο τη ε, επικεφαλή αντιπροσωπεία, επικεφαλή τη ε, υπηρεσία επίση που είναι υπεύθυνη για τα ζητήματα αυτά. Σα δίνουμε το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσά και την Επιτροπή στο σύνολό τη, γιατί ε, μα δώσατε, σε, δίνετε την ευκαιρία στι τελικέ αρχέ να μιλήσουμε για την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σας υπενθυμίζω ότι στο τέλος Δεκεμβρίου, στις 30 Δεκεμβρίου, ενακρίθη ένα ε, διάταγμα ε, το οποίο στην ουσία θέτει τέρμα ε, στην επίγουσα διαχείριση και στην έκτακτη διαχείριση της κατάστασης και ε, επαναφέρει την κατάσταση στην ομαλή διαχείριση και αναλαμβάνουν πάλι οι τοπικές αρχές. Ε, δηλαδή, να σας πω το εξής. Σήμερα η, η αντιπροσωπεία μας ε, αποτελείται αφενός μεν από συναδέλφου τη περιοχή τη περιφέρειας τη Καμπανία και αφετέρου από τους ανθρώπους ε, της ε, ε έκτακτης ομάδας ε, που ασχολήθηκε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τη διαχείριση για να σας δώσουμε κάθε δυσαφήνιση και κάθε απάντηση στα τυχόν ερωτήματά σας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε ε, να απαντήσουμε στις ανησυχίες ε, που δημιουργήθηκαν μετά από τις αναφορές ε, που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σας. Αν συμφωνείτε, να δώσω πρώτα το λόγο στο, στους συναδέλφους περιφέρειας της Καμπανίας και συγκεκριμένα στον κύριο Σατακρότη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, το πιο σημαντικό θέμα είναι ότι η περιφερειακή κυβέρνηση, οι περιφερειακές αρχές, ανακτούν εκ νέου όλες τις αρμοδιότητές τους μετά από μια μακρά περίοδο που είχε αναλάβει την διαχείριση η Ειδική Επιτροπή. Δημιουργούμε αυτή τη στιγμή ένα πλαίσιο για να επανέλθουμε στα συνηθισμένα μας, στην συνηθισμένη τάξη πραγμάτων. Η περιφέρεια πρόσφατα, το 2007 και 2008, απέκτησε περιφερειακούς νόμους που αναδιοργάνωσαν το πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων. Το πρώτο πράγμα που είναι σημαντικό γιατί αποτελεί και αντικείμενο μιας διαδικασίας επί παραβάση, είναι ότι κατά τη διάρκεια της περίοδου που είχε αναλάβει τα ενία η Ειδική Επιτροπή, είχε προβλεφθεί ένα νέο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο εφαρμόστηκε και ενσωματώθηκε από την περιφέρεια αλλά είμαστε ακόμη σε φάση έτσι βελτίωσης και τελειοποίησης του, ούτως ώστε να αποκτήσει η περιφέρεια ε, ένα μηχανισμό σχεδιασμού απόλυτα αναγκαίο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Τώρα, το ίδιο και για το σχέδιο διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων. Προβλέπετε προβλέπονται πάλι σχετικοί περιφερειακοί νόμοι και οι περιφερειακές αρχές έχουν εξοδοτήσει την ε, υπηρεσία για την ε, περιβαλλοντική προστασία της περιοχής, την άσπα. Να ασχοληθεί λοιπόν με αυτό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο πέρασε μετά από μια δημόσια πρώτη φάση συζήτησης σε μια δεύτερη φάση προετοιμασίας της περιβαλλοντικής έκθεσης, ούτως ώστε να εγκριθεί αυτή από τα όργανα συνδιαλλαγής. Δουλεύουμε λοιπόν και σε επίπεδο σχεδιασμού της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων αλλά και της διαχείρισης των ειδικών αποβλήτων. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι χάρη στα όσα προβλέπει το διάταγμα της κυβέρνησης υπήρξε μια επιτάχυνση του, των περιφερειακών νόμων και κανόνων με σκοπό τη δημιουργία επαρχιακών αρχών υπό τη μορφή εταιριών που θα έχουν καθήκον και να σχεδιάσουν με τη σειρά τους σε επίπεδο επαρχίας και να διαχειριστούν τον κύκλο των αστικών αποβλήτων. Θα έχουμε λοιπόν, φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή αυτό το δίκτυο των εταιριών και σιγά σιγά εντάσσονται στους παλιούς οργανισμούς που είχαν προβλεφθεί από ένα προηγούμενο νόμο του 1993, και οργανώνονται σε επαρχιακό επίπεδο για να διαχειριστεί σωστά ο κύκλος των αποβλήτων. Αυτές οι επαρχιακές ε, εταιρείε ξεκινούν με ένα προϋπολογισμό ο οποίος κληροδοτείται ε, από τη δομή της ε, Επιτροπής. Κατά την περίοδο που <clears throat> διαχειριζόταν, που διαχειριζόταν τα σκουπίδια αυτή η Επιτροπή, είχε προβλεφθεί ότι θα πρέπει να γίνεται η αποκομιδή των σκουπιδιών ανάλογα με το είδος. Θα πρέπει μάλλον να γίνεται μια πιο σωστή ανακύκλωση, ε, μια ανάκτηση ή τελικά αποκομιδή, διάθεση. Σε ό,τι αφορά την ανάκτηση. Υπάρχει αυτή η δομή της ε, Επιτροπής που προωθεί δράσεις ε, ενημέρωση, συντονισμού επαφών με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, που είναι και η παραγωγή αλλά και οι καταναλωτές, και έχουν αυξηθεί δραστηριότητες περί των σκουπιδιών ανάλογα με το είδος τους. Και έχουν εμπλακεί και διάφορες εταιρείες ε, συσκευασίας σε αυτόν τον τρόπο περισυλλογής ανάλογα με το είδος των σκουπιδιών. Επίσης, δίδονται χρήματα στις ε, κοινότητες, στους δήμους και στις κοινότητες, για να ενεργοποιήσουν και αυτές με τη σειρά τους ε, τα σχέδια ε, εξειδικευμένης περισυλλογής. Επίσης, δόθηκαν χρήματα για να αποκτηθούν ε, οι κατάλληλοι εξοπλισμοί, ούτως ώστε να γίνεται αυτή η εξειδικευμένη περισυλλογή των ε, απορριμμάτων ανάλογα με το είδος τους. Αυτά είναι τα οικονομικά στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σας πω ότι αυτή η δραστηριότητα δεν περιορίστηκε σε επίπεδο κυβέρνηση και περιφερειακών αρχών. Δεν περιορίστηκε λοιπόν σε μια μεταφορά κονδυλίων κοινοτικών από το προς, ε, τους Δήμους και τις κοινότητες για να προωθηθεί αυτό το, η προσπάθεια εξειδικευμένης περισυλλογής. Αλλά εντάχθηκε σε ένα πιο περίπλοκο, πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο που προβλέπει ότι από τον δημόσιο κορβανά θα προβλεφθούν κονδύλια για να πάνε στους Δήμους και στις κοινότητες, πέρα τα κοινοτικά. Και ενεκρίθη ένα πρόγραμμα, στα πλαίσια του οποίου η κυβέρνηση ίδια στηρίζει την περιοχή. Με στόχους συγκεκριμένους για τα απορρίμματα και με αυτό το σύστημα εμείς θα πολλαπλασιάσουμε τη χρηματοδότηση, δηλαδή πέρα από την κοινωτική χρηματοδότηση θα υπάρξει και μια εθνική. Μέσω αυτών των, ε, της εθνικής ε, χρηματοδότησης θα επιβραβεύσουμε τις κοινότητες και τους δήμους που θα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα ε, σε ό,τι αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών. Ε, πρόκειται για κάποια premium τα οποία θα δοθούν ε, είτε στις ε, περιφερειακές αρχές είτε στις τοπικές αρχές ανάλογα με τα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, μιλήσαμε για τα νομοθετικά στοιχεία, μιλήσαμε για τα οικονομικά στοιχεία. Δεν πρέπει να μιλήσουμε και το θέμα της παρακολούθησης. Η περιφέρεια έχει αποκτήσει ένα μέσο, ένα εργαλείο εντελώς καινούριο, μηχανοργανωμένο, που ονομάζεται παρατηρητήριο των απορριμμάτων και για τα αστικά απόβλητα χρησιμοποιήθηκε και από την Ειδική Επιτροπή για τη διαχείριση των, απο, των αποβλήτων. Υπάρχει δηλαδή μια τράπεζα δεδομένων που συλλέγει σε μηνιαία βάση και επεξεργάζεται τα ποσοστά αποκομιδής, εξειδικευμένης αποκομιδής, ανάλογα με το είδος των απορριμμάτων, ανακοινότητα. σε, κατά μέσο όρο, χάρη σε όλα αυτά τα μέτρα που σας περιέγραψα πριν, έφτασε και ξεπέρασε το μέσο όρο, η εξειδικευμένη εννοώ το 22%. Ε, φυσικά, ορισμένες τοπικές αρχές ε, έδειξαν υπερβάλλοντα ζήλο και ξεπέρασαν αυτό το ποσοστό. Ήταν πιο οργανωμένες και είχαν και μεγαλύτερες δυνατότητες, ε, γιατί είχαν καλύτερες εγκαταστάσεις ή περισσότερες εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της ειδική Επιτροπής χτίστηκαν, κατασκευάστηκαν φτιάχτηκαν μάλλον ε, αυτές οι επαρχιακές ε, εταιρείες οι οποίες ξεκινούν με ένα κεφάλαιο που τους ε, επιτρέπουν ήδη να είναι λειτουργικές από σήμερα. Ανέκτησαν επίσης όλο τον εξοπλισμό των προηγούμενων ε, και προϋπαρχόντων των φορέων, των φορέων που διαχειριζόταν τα, την αποκομιδή των απορριμμάτων. Τώρα, για να αποφασίσουμε ε, ποιος ε, διαχείριζεται καλύτερα τα απόβλητα. Θα, ε, έχουμε κάποιους δείκτες, ας πούμε πόσο, ποια κοινότητα έχει μεγαλύτερο ποσοστό αποκομιδής οργανικών απορριμμάτων. Χάρη στα κοινωνικά στην κοινωνική χρηματοδότηση ε, χρηματοδοτήσαμε και την επεξεργασία των απορριμμάτων, τόσο ώστε να μειωθεί η υγρασία ε, που εμπεριέχουν τα απορρίμματα αυτά, τα οποία πηγαίνουν, καταλήγουν τελικά στην χωματερή. Επίσης κάποια από αυτά, χάρη στην κοινωνική χρηματοδότηση, γίνονται κόμποστ. Κοπρόχωμα. τεχνητή κόπρος. Επίσης, ε, χάρη σε ένα πιλωτικό σύστημα, προσπαθούμε να κάνουμε μια ιχνηλασία των απορριμμάτων. Το Ιταλικό Υπουργείο ξεκίνησε με ένα σύστημα ιχνηλασίας των βιομηχανικών αποβλήτων. Και τώρα ε, στην περιφέρεια της Καμπανίας αυτό το σύστημα ανιχνευσιμότητας σε πειραματική βάση θα, θα συμπεριλάβει και τα αστικά απόβλητα. Δηλαδή θα υπάρξει δυνατότητα παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της ε, ε, ε, ε πορείας των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αρκούν αυτά τα οποία είπαμε ως ε, ένα γενικό πλαίσιο για να πούμε τελικά ε, και να τονίσουμε αυτό το οποίο γίνεται, ότι δηλαδή η περιφέρεια φεύγει από αυτή την, ε, την, έκτακτη ανάγκη. Κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να σας το αναφέρω είναι ότι στο νόμο πλαίσιο όχι, συγγνώμη λέει ο μιλητής, στον περιφερειακό νόμο προβλέπεται η σύσταση μιας ε, συγκεκριμένης ε, διεύθυνσης που θα ασχολείται με τα απόβλητα. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία φέτος και έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής αυτή τη υπηρεσίας. Ελπίζω λοιπόν όλες μας οι προσπάθειες να μας οδηγήσουν σε, σε, σε στα επιθυμητά αποτελέσματα. Λοιπόν, ευχαριστώ και σε αυτό το στάδιο διακόπτη πρόεδρο. Ρομπέρτο, Άνταμ, ο καθηγητής ε, κύριος Άνταμ θα έχει το λόγο εκ ε, αν συμφωνείτε, να δώσω το λόγο στον επικεφαλή της τεχνικής ε, ε υπηρεσίας, γιατί ε, θα μπορούσαμε με αυτόν τον τρόπο να, δω, να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Έχουμε τον κύριο Φιλιορία, τώρα, ο οποίο είναι νομικός ε, και ο οποίο είναι επικεφαλή τη τεχνική υπηρεσία του Υπουργού Μπερτολάζου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα ακούσαμε τι ε, απόψει. Ε, της ε, περιφέρειας όλων των υπηρεσιών, όλα αυτά που κάναμε για να φύγουμε από αυτή την έκτακτη ανάγκη, μετά από 15 χρόνια μια ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, πραγματικά φτάσαμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Με το διάταγμα ε, του Μαΐου του 2008, οι στόχοι οι οποίοι είχαν αναφερθεί και είχαν εντοπιστεί, ήταν να φύγουμε την 31η του ε, Δεκεμβρίου 2009 από αυτή την κατάσταση που όπως σας είπα διαρκούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από την άλλη να υπάρξουν οι επαρκείς υποδομές στην περιφέρεια έτσι ώστε να είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αυτή η συγκεκριμένη ανάγκη. Η διαχείριση δηλαδή του κύκλου των απορριμμάτων στην περιοχή της Καμπανίας. Αυτή η στόχη επιτεύχθηκαν επιτεύχθηκαν μέσω πολλών πρωτοβουλειών. Η πρώτη και ίσως και η πιο σημαντική ήταν η πραγματοποίηση πολυάριθμων χώρων υγειονομικής ταφής ε, μετά από συγκεκριμένα ε, ε, νομικά, νομοθετικά διατάγματα, σεβόμενοι απόλυτα την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, χώροι υγειονομικής ταφής που σίγουρα μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να μιλήσουμε για μια αυτονομία τη περιφέρεια τη Καμπανία μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Καμπανία από άποψη υποδομή ε, είναι πρότυπο για τη χώρα, υπόδειγμα. Ίσως είναι η περιφέρεια με την περισσότερη υποδομή και την καλύτερη υποδομή. Ε, υπάρχουν εγκαταστάσεις διαλογής ε, ε, εγκαταστάσεις οι οποίες είναι πολύ καλές, εξυγχρονισμένες, επαρκείς. Έχουν, υπάρχουν ακόμα διαδικασίες βελτίωσης με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι ε, πριν διατεθούν οριστικά τα απορρίμματα, έχουν αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης και διαλογής για, με στόχο την καλύτερη προστασία ε, της, ε, των κατοίκων της περιοχής. Πριν δηλαδή ε, πάνε στο τελικό τους προορισμό τα απόβλητα. Το διάταγμα διευκρινίζει συγκεκριμένα το πού θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις και αυτό ε, μέσω μιας ολοκληρωμένης έρευνας που, θα επρεπε να πραγματοποιηθουν αυτες οι εγκαταστασεις και αυτο μεσω μιας ολοκληρωμενης ερευνας που ελα που και εκεί ελήφθησαν υπόψη όλα τα συμφέροντα που μερικές φορές ήταν και αντικρουόμενα με στόχο την εξασφάλιση της ορθής διαχείρισης του κύκλου των αποβλήτων. Αυτή η διαδικασία βεβαίως συνοδεύτηκε με την ε, τεχνολογική εξέλιξη, με το χώρο της ατσέρα αξιοποίησης ε, για των αποβλήτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ε, που σήμερα μπορούμε να πούμε ότι περίπου 2.000 τόνους την ημέρα, επεξεργάζεται υλικό 2.000 τόνους την ημέρα. Και για να καταλάβετε το πόσο σημαντική είναι αυτή η εγκατάσταση, αρκεί να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μέση παραγωγή που είναι κάτω από τις 5.500 τόνους το την ημέρα ε, ε, απόβλητα, έτσι. Αυτή λοιπόν η εγκατάσταση στην Ατσέρα, που μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές, να μην σας πω η πιο σημαντική εγκατάσταση σε όλη την Ευρώπη, μπορεί να απορροφήσει, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ρήμα απορροφήσει, σχεδόν το 40% της, ε, παραγωγή, της ημερήσιας παραγωγής αποβλήτων στην περιφέρεια. μία εγκατάσταση που να σας πω ότι ε, είναι το καμάρι μας κατά κάποιο τρόπο. Γιατί μιλάμε για μια εγκατάσταση που αποτεφρώνει τόσο, σημαντικά, ε, ε, τόσο σημαντικές ποσότητες αποβλήτων και μας έδωσε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ε, τις, ε, τις, τις προβλεπόμενες επιδόσεις του σχεδίου αυτού. Όχι μόνο η εγκατάσταση αυτή σέβεται απόλυτα την κοινοτική νομοθεσία, αλλά σέβεται ε, ένα ειδικό ε, περιβαλλοντολογικό πλαίσιο νομοθετικό, το οποίο ορίστηκε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και σε όλες τις λεπτομέρειες και που αφορά την συγκεκριμένη κατάσταση και, και τα, ε, οι προδιαγραφές είναι πολύ πιο αυστηρές από αυτές που προβλέπει η εθνική και η κοινωτική νομοθεσία. Αν θεωρείτε σκόπιμο, μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τα λεγόμενά μου. πέραν των πολεμικών επικρίσεων που ακούστηκαν μερικές φορές, ε, ε, να σας πω ότι τα στοιχεία όχι μόνο μας καθησυχάζουν, αλλά είναι τέτοια που ε, οδήγησαν την κυβέρνηση στο να υλοποιήσει όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να μπορέσει η περιφέρεια της Καμπανίας να είναι προσαρμοσμένη απόλυτα σε απαιτήσει επεξεργασίας του κύκλου των αποβλήτων και να φτιάξουμε και άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από τα απόβλητα. Όχι μόνο παράγουν ενέργεια, αλλά διοχετεύουν ε, τα, τα απορρίμματα με απόλυτη ασφάλεια. Η τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας μας έχει οδηγήσει σε τρομερά αποτελέσματα. Και ε, από τώρα μπορούμε να σας πούμε, παρόλο που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες, ότι όχι μόνο έχουμε επίτευξη των αρχικών στόχων του σχεδίου, αλλά το 20-25% περίπου οι εκπομπές είναι στο 20-25% του, ε, του συνολικού ε, ποσού εκπομπών όπως αναφέρει στην νομοθεσία. Δηλαδή βρισκόμαστε πολύ πιο κάτω. Ε, Λοιπόν, όσον αφορά τι ε, εγκαταστάσει αυτέ, μπορώ να σα πω ότι τα αποτελέσματα μα οδηγούν στο εξή συμπέρασμα. Θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η εγκατάσταση ε, ε, μέσα σε απόλυτη συμφωνία με τον νόμο. Σημαντική ήταν η όθηση που εδόθη για την ε, διαλογή των απορριμμάτων. Όπως είπε και πριν από λίγο ο εκπρόσωπος της Καμπανία, ε, διπλασιάσαμε ε, αυτά τα οποία κάναμε σε, ε, αυτά, ε, σε επίπεδο διαλογής σε σχέση με τα αυτά που κάναμε πριν από 1,5 χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τελικά ε, τα απόβλητα τα οποία πηγαίνουν στους χώρους υγειονομικής ταφής είναι πολύ λιγότερα. Δηλαδή, ξεχωρίζουμε και διαλέγουμε τα απόβλητα με αποτέλεσμα ε, να έχουμε αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Σε σχέση με αυτά τα θετικά, τη θετική εικόνα, που ήταν το αποτέλεσμα σκληρής εργασία για 1,5 χρόνο περίπου. Και θα σας έλεγα, σε απόλυτη συμφωνία ε, και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση συμμετείχε ε, και ε, η δομή της ε, πολιτικής προστασίας και αντίστοιχες υπηρεσίες και, και υπήρξε απόλυτη συμφωνία, όπως σας είπα, με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πάντα ήταν κοινή η στόχη και είχαμε και συμβολή μέσω know-how δηλαδή. Ε, μέσω συγκεκριμένη τεχνογνωσία. Δηλαδή ε, ε, η τοπική αυτοδιοίκηση βοήθησε τις προσπάθειες της Ε, των εθνικών αρχών. Και επειδή τελειώνει τώρα, τέλειωσε αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προχωρήσαμε στο ροντάρισμα, αν θέλετε, της κατάστασης που θα ακολουθήσει μετά την επίγουσα και έκτακτη ανάγκη. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναλάβει μία ε, ε, συντονισμένη δράση για να δούμε το πώς όλες αυτές οι γνώσεις, η τεχνογνωσία, οι τεχνικές που εφαρμόσαμε αυτά τα χρόνια, πώς μπορούν τώρα να κληροδοτηθούν στην περιφέρεια για να μπορέσουμε να ε, πλαισιώσουμε καλύτερα αυτέ τι πρωτοβουλίε και τι τωρινέ αλλά και τι ε, μελλοντικέ, αυτέ που θα δώσει ω απάντηση η αυτοδιοίκηση στα προβλήματα που θα δημιουργηθούν σε αυτό το τόσο λεπτό και δύσκολο θέμα. Προβλέψαμε λοιπόν μια περίοδο, ένα χρονικό διάστημα, όπου η κεντρική διοίκηση θα εξακολουθήσει να ασκεί ε, τις, ε, ε, συγκεκριμένη δράση, δράση συμβούλου, δράση υποστήριξης και αρρωγής και συνδρομής των τοπικών αρχών, που σίγουρα αναλαμβάνουν το δύσκολο καθήκον να επανενταχθούν με βάση τη συγκεκριμένη νομοθεσία ε, ε, σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο και να λάβουν τα καθήκοντά τους. Επίσης, όπως ε, γνωρίζετε, προβλέπουμε ε, και εφαρμογή συστήματος κυρώσεων. Με το νομοθετικό διάταγμα 172-2008 η κυβέρνηση θεώρησε σκόπιμο να ε, σκληρύνει τη στάση της και σε επίπεδο κυρώσεων, διοικητικών κυρώσεων, αλλά και σε επίπεδο ποινικό έναντι των παραβατών σε αυτό το τόσο δύσκολο ζήτημα. Όσον αφορά αυτό το σύστημα, το ε, ε, ιδιαίτερα αυστηρό σύστημα κυρώσεων, πρέπει να πω ότι ε, η, η κοινότητα συνολικά απάντησε θετικά, ανταποκρίθηκε σχετικά. Βεβαίω, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά ε, σήμαιναν ότι έπρεπε να αλλάξει κοινοτροπία. Και βέβαια, ε, έχουμε τώρα και πολύ μεγαλύτερα ποσοστά διαλογή, το είπαμε ήδη. Και θα, ε, αυτό δεν θα μπορούσε να έχει γίνει χωρίς την ε, αμέριστη ε, συνεργασία των πολιτών. Και από την άλλη Έχουμε λοιπόν τη συνεργασία των πολιτών και από την άλλη τις κυρώσεις που έχουν ως στόχο να οδηγήσουν στην άμεση πάυση παράνομων δραστηριοτήτων και την αποφυγή νέων τέτοιων πράξεων στο μέλλον πολύπλοκο το σύστημα, διαρθρωμένο σύστημα, το οποίο δομημένο σύστημα που οδήγησε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην νομοθεσία που θα εγκριθεί το 2010. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή κατά την άποψή μας πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις και θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να ομαλοποιηθεί απόλυτα η κατάσταση. Βεβαίω, η Ιταλική κυβέρνηση ε, μπορεί να σας δώσει περαιτέρω συμπληρωματικά στοιχεία για να μπορέσετε όλοι να καταλάβετε και να επαληθεύσετε αυτά τα οποία σας αναφέραμε ως αποτελέσματα και όσον αφορά ε, τις ικανότητες, τις περιφέρειες για να, μην, για να αποτρέψουμε τελείως μία επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Perfetto. Allora passo la parola al rappresentante della Commissione. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα και εγώ να παρέμβω για τις αναφορές που βρίσκονται στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Αναφορές τις οποίες έχουμε ήδη συζητήσει και κατά τις οποίες η Κομισιόν σε μια προηγούμενη συνεδρίαση στην 1 την 1η Δεκεμβρίου του 2009 είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει την άποψή τους την άποψή της. Επομένως, δεν πρόκειται να καθυστερήσω τα μέλη της Επιτροπής σας, επαναλαμβάνοντας τα όσα είχα πει την 1η Δεκεμβρίου. Πριν παρουσιάσω τα δύο σημεία που αποτελούν το αντικείμενο της ε, προσφυγής μας ε, στο ΔΕΚ και το θέμα των, χρηματικών, ε, των χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέμα του οποίου ζητήθηκαν πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τις Ιταλικές Αρχές που μας έδωσαν κάποιες πληροφορίες όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που ξεκίνησε η διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής και Ιταλικής Κυβέρνησης για τη διαχείριση των ε, αποβλήτων στην Καμπανία. Πολλές φορές ζητήσαμε από τις Ιταλικές Αρχές να μας ενημερώσουν και οι σημερινές προφορικές πληροφορίες είναι οι πρώτες ουσιαστικά πληροφορίες που λάβαμε για τη σημερινή κατάσταση, για την τρέχουσα κατάσταση. Η διαδικασία επιπαραβάση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2007 για παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν συνεχεία έλαβε την απόφαση να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον Μάιο του 2008 και η ακρόαση, η ακροαματική διαδικασία στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου έγινε στις 3 Δεκεμβρίου του 2009, δηλαδή δύο μέρες μετά τη συνεδρίαση όπου συζητήσαμε τις ιταλικές αυτές αναφορές. Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η απόφαση θα ληφθεί χωρίς αναμονή και χωρίς να περιμένουμε τα συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέα. Προφανώς, εγώ από πλευράς Κομισιόν δεν μπορώ να σας δώσω ενδείξεις για την ημερομηνία της κραματικής διαδικασίας, της απόφασης, αλλά πιστεύουμε ότι η απόφαση θα έχει εκδοθεί πριν το καλοκαίρι τους επόμενους μήνες κατά πάσα πιθανότητα. Κατά την άποψη της Επιτροπής, με την υιοθέτηση ενός χρονοδιαγράμματος και την εφαρμογή, καθώς και την υλοποίηση διαφόρων υποδομών για την διάθεση των αποβλήτων. Όλα αυτά είναι στοιχεία μιας ε, συνεπούς διαχείρισης της ε, διάθεσης των αποβλήτων και θα επιτρέψουν σίγουρα στην ε, καμπανία να, υιοθετηθεί με να υιοθετήσει συγγνώμη, ένα νομοθετικό πλαίσιο για να ευθυγραμμιστεί με τα όσα επιτάσσει η κοινοτική νομοθεσία. αν ε, το δικαστήριο αποφασίσει υπέρ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποφασίσει ότι παραβιάστηκε το κοινοτικό ε, δίκαιο, Αν αποφασίσετε, συγγνώμη, ότι παραβιάσετε το κοινοτικό δίκαιο, τότε σημαίνει ότι το δικαστήριο αποφασίζει υπέρ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά την κρίση που έγινε που παρουσιάστηκε το 2007 σε αρχές της Άνοιξης, η συγχρηματοδότηση στον τομέα των αποβλήτων και μόνο σε αυτόν σταμάτησε για την καμπανία από τον Ιούνιο του 2007 και μετά. Οι πληρωμές οι οποίες έχουν γίνει αφορούν τις περιόδους 2000, 2006, 2007, 2013. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η απουσία ενός κατάλληλου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή που αποτέλεσε τη βάση για την διαδικασία που διαπιστώθηκε, παράβαση που διαπιστώθηκε από την ε, Κομισιόν και που αποτελεί παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας εν προκειμένου, δεν έδινε τις απαραίτητες εγγυήσεις για τη σωστή χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων. Και γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν αναγκάστηκε να μπλοκάρει την χρηματοδότηση. Η Ιταλία έκανε δύο προσφυγές σε πρωτοβάθμιο δικαστήριο εναντίον της απόφασης της Κομισιόν να σταματήσει τη συγχρηματοδότηση για την περίοδο 2000-2006. Και αυτές οι προσφυγές εκρεμούν ακόμα, δεν έχουν εκδικαστεί. Εξυπακούεται ότι η Κομισιόν μπορεί να αναθεωρήσει την απόφαση άρσης της συγχρηματοδότησης, αναστολής της συγχρηματοδότησης, όταν η κατάσταση στην καμπανία αλλάξει. Και αυτό πιστοποιηθεί από στοιχεία. Τα βασικά στοιχεία για να ενεργοποιηθεί εκ νέου η χρηματοδότηση, η συγχρηματοδότηση θα είναι ο καθορισμός ενός προγραμματισμού στον τομέα αυτό μέσω ενός προγράμματος διαχείρισης των αποβλήτων που θα συμπεριλαμβάνει ένα κατάλληλο δίκτυο υποδομών διάθεσης από τη μία των αποβλήτων, τελικής διάθεσης και όλα αυτά με μία λογοδοσία ε, που θα βασίζεται σε γεγονότα, σε ντοκουμέντα, σε στοιχεία. Από την άλλη πρέπει να βγει η καμπανία από το ειδικό καθεστώς της ειδική Επιτροπής και να επανέλθει σε μια συνηθισμένη διαχείριση, καθημερινή διαχείριση των αποβλήτων. Να ξεφύγει λοιπόν από το ειδικό καθεστώς της Επιτροπής. Και αν κατάλαβα καλά από τις παρουσιάσεις, ε, προς αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε. Θα ήθελα να επαναλάβω κάτι που αφορά τις αναφορές. Ότι εμείς ως Επιτροπή δεν έχουμε την αρμοδιότητα να παρέμβουμε στις αποφάσεις των κρατών μελών. Αποφάσεις για τις νέες εγκαταστάσεις διάθεσης των αποβλήτων. Δεν έχουμε εξουσία για να αποφασίσουμε πού θα τοποθετηθούν τα διάφορα εργοστάσια, οι διάφορες εγκαταστάσεις. Απλώς θέλουμε ολόκληρο το πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου να γίνει σεβαστό. Ευχαριστώ κυρία Σαπουτσέλα. Τώρα θα ξεκινήσει η συζήτηση η κυρία Μέρκες. Uh, thank you, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και τις Ιταλικές Αρχές για την έλευσή τους εδώ και τις εξηγήσεις που έδωσαν μου παραμένουν ανοιχτά ορισμένα ερωτηματικά, διότι ομολογώ ότι οι ανησυχίες μου δεν καλύφθηκαν όλες. Για παράδειγμα, ακούω ότι η καμπανία έχει όλων των ειδών νέες εγκαταστάσεις και μάλιστα θα γίνει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Τι γίνεται όμως με τις παλαιές εγκαταστάσεις. Αυτές συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα από την κοινοτική νομοθεσία. Υπάρχουν ορισμένε νέε εγκαταστάσει, αλλά υπάρχουν και παλές εκατοντάδε, οι οποίες ε, δεν είναι σύμμορφε με την ε, ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τότε το πρόβλημα παραμένει. Ακούω ύστερα για πολλές πρωτοβουλίες, καλέ πρωτοβουλίες αυτές, και βλέπω ότι υπάρχει καλή θέληση για να επιληθεί αυτή, αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Πολλές πρωτοβουλίες όμως αυτομάτως θέτουν το ερώτημα ποιο ασκεί τον συντονισμό. Αυτές οι πρωτοβουλίε συντονίζονται από κάποιον και ποιο ασκεί τον συντονισμό. Ακούσαμε τους αναφερομένους και σε ό,τι τους αφορά υπάρχουν αρχές, οι αρχές όμω δεν είναι καλά συντονισμένες. Δεν άκουσα και τι γίνεται με την υγεία. Μιλήσατε πολύ για υποδομές, για νέες εγκαταστάσεις για την ε, κατανομή των απορριμμάτων, αλλά τι γίνεται με την υγεία. Έγιναν εξετάσεις, έγιναν εξετάσεις μάλλον και έδειξαν ότι η κατάσταση είναι πολύ άσχημη. έχουν γίνει νέες εξετάσεις που έδειξαν εν τέλει ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας των ε, πολιτών. Uh, uh, Εγώ εκπλήσωμαι. Μου φαίνεται ότι εν τέλει καίνε όλα τα σκουπίδια στην περιφέρεια αυτή. Δεν είναι και η καλύτερη λύση. Ίσως είναι βέβαια σύμμορφη με την οδηγία περί απορριμμάτων. Αυτή όμως η ίδια η οδηγία είναι ασθενείς, είναι αδύναμη, Άρα δεν παραβιάζεται μεν η οδηγία, αλλά δεν είναι σύγχρονη και καλή λύση. Είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς να καίει τα σκουπίδια. Το τελευταίο πράγμα. Και εδώ μου λέτε ότι είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε. Συνδέω εδώ και μια ερώτηση προς την Επιτροπή, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τουλάχιστον να μην το χρησιμοποιήσετε ως ανανεώσιμη ενέργεια. Να μην χρησιμοποιούν χρήματα για τις ανανεώσιμες για αυτό το πράγμα που είναι μια πραγματικά πρωτόγονη μορφή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επίσης πρωτόγονη ε, μορφή διαχείρισης του προβλήματος των απορριμμάτων. Και είπατε 22% είναι πάρα πολύ χαμηλό. Και είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, διότι αν υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα τότε παραβιάζεται παντός είδους κανόνες και είναι και κοντά σε αστικό κέντρο. Η ερώτησή μου τώρα προς τις Ιταλικές αρχές. Θεωρείτε την καύση σύγχρονο τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων και μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι στα απορρίμματα που καίτε εν τέλει δεν περιλαμβάνονται και επικίνδυνες ουσίες και με ποιο τρόπο το ελέγχετε. Εμείς, ε, εγώ είμαι Δανέζα και στη Δανία έχουμε πολλά προβλήματα με διοξίνες αν και έχουμε μάλιστα και ένα ε, πάρα πολύ προηγμένα συστήματα καύσης. Παρ' όλα αυτά έχουμε πάρα πολύ δυσκολίες. Εκπλήσωμε. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την επεξεργασία της αναφοράς, διότι τη λυπάμαι πραγματικά αυτή την περιφέρεια. Δεν μου φαίνεται να έχουν λυθεί τα προβλήματα, αλλά απλώς κάπως έχουν εμβαλωματικά αντιμετωπιστεί. Ε, Θέλουν ε, οι αναφέροντες να παρέμβουν πάρα πολύ σύντομα, γιατί θέλουν να κάνουν κάποιες διευκρινήσεις. Κοιτάξτε, επειδή έχει, βεβαίως έχει περάσει η ώρα, αλλά σας παρακαλώ, μόνο ένας ε, να μιλήσει εξ ονόματος όλων σας και όχι πάνω από δύο λεπτά. Αν ε, μου δίνετε την άδεια, να δώσουμε τη δυνατότητα και στους αναφέροντες να απαντήσουν. Μάλιστα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Εξ ονόματος και των υπολείπων αναφέροντων. Δεν θέλω να σας κλέψω το χρόνο. Μιλάω για όλες τις αναφορές που κατατέθηκαν. Από αυτούς τους πολίτες του Τζουλιάνο, της Ατζέρα και των άλλων κοινοτήτων. Εδώ δεν θα μιλήσουμε για τους λόγους που μας οδήγησαν στα παράπονα. Αλλά θέλω να απαντήσω ε, για αυτά που ακούσαμε. Και μετά από αυτά που είπε η Κομισιόν πρέπει να γίνουν κάποια, κάποιοι σχολιασμοί. Η κυρία Πουτσέλα. Νομίζω ότι αναγνωρίζουν την προσπάθεια που έκαναν αυτούς τους μήνες και αυτά τα χρόνια οι αναφέροντες. Γιατί με, την τελευταία, με το τελευταίο διάταγμα, νομοθετικό διάταγμα, πρέπει να σας πω κάτι δυσάρεστο. Ε, ακούσαμε κάποια πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω ότι τα αντίθετα έχουν ε, συμβεί. Στην πραγματικότητα δεν βγαίνουμε από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην καμπανία σε ό,τι αφορά την διαχείριση των σκουπιδιών. Δεν ε, πλησιάζουμε στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ε, αναγνωρίστηκε ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά η οδηγία 2006 12. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είπε ότι δεν υπάρχει υποδομή για τη διάθεση των σκουπιδιών. Ε, όμως, στο μεταξύ υπάρχει νέα οδηγία του 19 της ε, του 2008. Στο άρθρο 4 ε, μιλάει για την ιεράρχηση των αποβλήτων. Ε, από αυτά που ακούσαμε, στην πραγματικότητα, ποια είναι η αρχή στην καμπανία, φτιάχνουμε απλώς πέντε αποτεφρωτές. Τίποτε άλλο. Ποια είναι η διαφοροποιημένη ε, περισυλλογή. Τίποτα δεν έχει γίνει. Με το νέο νομοθετικό διάταγμα επίσης ε, το οποίο εγκρίθηκε δεν απαντάμε καθόλου συγκεκριμένα πώς γίνεται η διάθεση των ε, αποβλήτων. Και το άρθρο 28 της νέας οδηγίας πλαίσιο επίσης, αυτό που μιλάει για ένα σχέδιο διάθεσης των αποβλήτων. Αυτός ο αποτεφρωτής της Ατζέρα είναι το μοναδικό πράγμα που υπάρχει. Ο κόστος αυτής, το κόστος αυτής της εγκατάστασης είναι 370 εκατομμύρια ευρώ.